Είναι μια πρωτοβουλία που θα χρειαστεί δύο διαδοχικές τρόικες να την ε, συνεχίσουν. Κύριε Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας θα οργανώσουμε στο και δύο υψηλού επίπεδου διασκέψεις σχετικές με την υγεία και βέβαια μεγάλος αριθμός συνεδριάσεων θα γίνει και σε τεχνικό επίπεδο. Η πρώτη υψηλού επίπεδου διάσκεψη ε, που ονομάζεται το Φόρουμ της Αργυράς Οικονομίας, Silver Economy Forum, ήδη έλαβε χώρα πριν από δύο εβδομάδες περίπου. Αναφέρθηκε σε ε, θέματα που αφορούν την γύρανση ε, ή μάλλον την ε, τρίτη ηλικία σε όρους υγείας και δραστηριότητας αλλά και τις αλλαγές ε, με τα νέα μακροοικονομική πραγματικότητα που συνεπιφέρει αλλά και την κοινωνική αναγνωρίστηκε ότι το να γυράσκει κανείς πρέπει να, ότι η γύρανση του πληθυσμού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην, στο κοινωνικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων αλλά και στις στρατηγικές για την επιχειρηματικότητα ε, γενικά ε, και έχουμε και τη δεύτερη διάσκεψη στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου για την οικονομία της ευημερία. Κύριε Πρόεδρε, συνολικά μπορώ να πω καταλήγοντας ότι οι μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες που προκύπτουν πολλές ε, στον ορίζοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετίζονται με αλλαγές που έχουν να κάνουν με την παγκοσμιοποίηση, την κλιματική αλλαγή, τη μετανάστευση, τεχνολογικές εξελίξεις, νέες μορφές εργασίας, γύρανση του πληθυσμού ή γυράσκοντες πληθυσμούς και την αύξηση της παραπληροφόρησης και όλο και ενισχυόμενη δυσπιστία σε σχέση με την επιστήμη που δείχνουν οι πολίτες. Ταυτόχρονα όμως τα συστήματα δημόσιας υγείας σε όλη την Ευρώπη δυσκολεύονται μεταξύ άλλων ε, να καλύψουν και το αυξημένο κόστος ή τις υψηλότερες απαιτήσει των ε, ασθενών, την τεχνολογική μετατροπή, την ε, έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, την δυσπιστή απέναντι στον εμβολιασμό ή άλλες προκλήσεις που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε φάρμακα. Ε, εν προκειμένου λοιπόν η ανθεκτικότητα αλλά και η ικανότητα για ταχεία προσαρμογή σε αλλαγέ σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας είναι όλο και περισσότερο σημαντικές. Προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτές ε, τις αλλαγές που προκαλούν αυτές οι μεγάλης κλίμακας εξελίξης, αλλά και να ε, εξασφαλιστεί ε, βιώσιμη και ανοιχτή προς όλους ε, ανάπτυξη, πρέπει να προαγάγουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Αυτό το κοινωνικό μοντέλο το οποίο γεννά σταθερότητα, το οποίο συνιστά ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην όλο και πιο δύσκολη, στο όλο και πιο δύσκολο περιβάλλον παγκόσμιου ανταγωνισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει να είναι όχι μόνο η πιο ανταγωνιστική, αλλά και η οικονομία με τη μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή στον κόσμο. Κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η κατεύθυνση, όπως σας την περιγράφω, η κατεύθυνση που θα θέλαμε να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα πέντε χρόνια. Η προσέγγιση που προτείνουμε, η οικονομία της ευημερίας, της ευημερίας είναι μόνο ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Ελπίζουμε να προσφέρουμε στις μελλοντικέ προεδρίες μια βάση, ένα γερό θεμέλιο πάνω στο οποίο να μπορούν να χτίσουν τις περαιτέρω τους δράσεις όπως αυτές χρειάζονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας αυτή. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στους συντονιστές των διάφορων πολιτικών ομάδων και θα αρχίσουμε με το ΕΛΚ. Πίτερ Λίζε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Αν θέλουμε να ευχηθούμε, να χαρούμε κάποιον, ε, να το ευχηθούμε για την γενέθλιά του ή καλή χρονιά, λέμε ε, δύναμη, ανάπτυξη, διαφάνεια, σημαντικά είναι αυτά. Αλλά τι λέμε κυρίως, υγεία, να είναι υγιής κάποιος, αυτό ευχόμαστε και το ίδιο ε, ισχύει για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Υγεία. Πρέπει να είναι μια προτεραιότητα φυσικά και σεβόμεθα τι συνθήκε και υπάρχουν κάποια ζητήματα που αποτελούν και αρμοδιότητα. Αλλά η συνθήκη μα δίνει και τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση εκεί όπου έχει αρμοδιότητα η Ευρώπη να πρέπει να λαμβάνει δράση σε ό,τι δεν αφορά ε, τον ε, μέχρι τώρα Επίτροπο της Υγείας. Ε, ήταν μια απογοήτευση η δράση του. Έκανε μια πρόταση, μετά το Συμβούλιο δεν άλλαζε θέσεις και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει πρόοδος. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα και πρέπει να την αδράξουμε με τη νέα ε, πρόεδρο της ε, Επιτροπής που είναι γιατρός στο επάγγελμα και νομίζω ότι καλό είναι να μπει εκεί εστίαση ε, στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Και θα πω ε, για δύο πράγματα, κυρίως για το καρκίνο. Ο Μάφρετ Βέμπερ, ο δικός μας κορυφαίος υποψήφιο, είχε βάλει στο επίκεντρο την αντιμετώπιση του καρκίνου και οι τέσσερις μεγάλες ομάδες το είχαμε συμφωνήσει γιατί θεωρούσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρώπη να υπάρξει βελτίωση στον αγώνα κατά του καρκίνου. Το δεύτερο θέμα που θέλω να ε, ζητήσω να στηρίξετε είναι η ατοχή ε, στα αντιβιωτικά και τα αντιμικροβιακά. 33.000 άνθρωποι χάνουν τον χρόνο τη ζωή του κάθε χρόνο με βάση τα στοιχεία της ε, CDC από την από στελέχη που είναι ανθεκτικά στα αντιβιωτικά ή στα αντιμικροβιακά φάρμακα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν ε, εξελίξεις. Θέλουμε καινοτομία, θέλουμε νέα φάρμακα αν δεν έχουν δράσει πλέον ε, τα ισχύοντα. Σίγουρα είναι η πρόληψη σημαντικό, αλλά αν πεθαίνει κόσμος θέλουμε και θεραπεία, θεραπείες να βρούμε και θέλουμε λοιπόν να έχουμε την υποστήριξή ώστε να έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση από την ε, πλευρά της Ευρωπαϊκή Ευχαριστούμε. Ε, εκ μέρους των σοσιαλιστών, ο κύριος Σε Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ, που ήρθατε. Είναι καλό που ακούμε ότι η πρόληψη βρίσκεται πάνω-πάνω στις προτεραιότητές σας όσον αφορά την προσέγγισή σας. Ρώτησα νωρίτερα και την Υπουργό Περιβάλλοντος και θα σας ρωτήσω το ίδιο για τα εμβόλια και το ότι οι άνθρωποι διστάζουν πολλές φορές να προβούν σε εμβολιασμό. Εμείς θα στηρίξουμε το δικαίωμα των γονιών να μην εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Θα μειώσουμε την πίεση πάνω στους γονείς να εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Εγώ δεν θα ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο. Φοβάμαι όμως γιατί υπάρχουν υπόνοιες για κάποιες πτυχές της επιστήμης που οδηγούν σε κακά αποτελέσματα. Αν δούμε το 30% που αυξήθηκε η λαρά και πόσες ασθένειες ξεσπούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μέτρα πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε για να υπάρξει συνένεση μεταξύ των χωρών μελών και να πιστέψει το κοινό και πάλι την επιστήμη ώστε να αυξηθεί η σιγουριά που νιώθει ο κόσμος για το ότι είναι καλά τα εμβόλια, για παράδειγμα. Και θα μπορούσε να υπάρχει ένα πρόγραμμα για ένα σύστημα έγκρισης εμβολιασμών, το οποίο υπάρχει βέβαια και είναι καλό, αλλά ίσως δεν είναι αρκετά γνωστό μεταξύ των πολιτών να μάθουν οι πολίτες ποια ακριβώ είναι η διαδικασία, δηλαδή να υπάρξει κάποιο ρόλος διαπαιδαγώγησης ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος και να μην ε, αντιδρά με υποψία απέναντι στην επιστήμη και τις αποφάσεις μας. Ευχαριστούμε, Βερονίκ Διελβιά, εκ μέρους του Ρινιού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ που μας παρουσιάσατε τα θέματα της υγείας και όχι μόνο τα αρνητικά, αλλά μια συνολική άποψη με πολύ αλληλεγγύη. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού που ονομάσατε εσείς η οικονομία της ευημαρίας, η πρόληψη δηλαδή των κινδύνων που έχουν να κάνουν με τα τρόφιμα και με το περιβάλλον, αυτά πράγματι θα πρέπει να μείνουν στο πυρήνα της ενασχόλησής μας εννοείται ότι είναι προνόμιο η υγεία των χωρών μελών. Όμως, τα θέματα η υγεία, όταν πρόκειται για υγεία μιας ολόκληρης κοινωνίας ή διαφόρων κλάδων, το είπατε κι εσείς, δεν λαμβάνονται δυστυχώς ακόμα αρκετά υπόψη, ούτε και το θέμα του καρκίνου και επανέρχομαι σε αυτό. Σκέφτομαι επίσης και τη γύρανση των πληθυσμών την ψηφιακή υγεία και την εξάπλωσή της, πώς επιστρέφει κανείς στη δουλειά του μετά από μακρόχρονη απουσία λόγω σοβαρής ασθάνειας. Και σκέφτομαι επίσης και την ψυχική υγεία και σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε σε αυτό. Σκέφτομαι επίσης και την αναπαραγωγική υγεία που απασχολεί πολύ τις γυναίκες ιδιαίτερα και που εμπίπτει επίσης στα πλαίσια αυτού που ονομάσατε εσείς ευημερία. Αυτά τα θέματα είναι πολλά και διάφορα και γι' αυτό πρέπει να δεσμευτεί το Συμβούλιο. Είναι... Πρέπει να δούμε τι θα κάνει η πρόεδρος της Επιτροπής. Δεν μπορούμε να φανταστούμε όλα αυτά να μην τα συνδέσει η με κάποιο τρόπο και ελπίζουμε η, εντολής, η εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι πιο δραστήρια από ό,τι ήταν η προηγούμενη. Όσον αφορά για την Προεδρία του Συμβουλίου, ε, περιμένουμε μια φιλόδοξη αντιμετώπιση και μέτρα που θα φροντίσουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές να έχουν πραγματικά θετική επίπτωση πάνω στους Ευρωπαίους πολίτες και στα παιδιά τους. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους των Πρασίμων τώρα, η κυρία Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ και σας ευχαριστούμε που ήρθατε και που μας παρουσιάσατε τους στόχους σας. Πραγματικά, πραγματικά εκτιμά όλους ιδιαίτερος την επιθυμία σας να προστατεύσετε την υγεία των πολιτών και κυρίως μου αρέσει πολύ αυτή η συνολική άποψη που έχετε και προσέγγιση για το θέμα. Θέλω όμως να επιστήσω την προσοχή σας ε, κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με την υγεία και την ευημερία των πολιτών. Και θέλω να ξέρω κατά πόσο ένα μη τοξικό περιβάλλον, αν για σας θα είναι ένα θέμα γιατί ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα δεν έχει προσφέρει μια στρατηγική για αυτό το θέμα, ενώ θα έπρεπε να ήταν έτοιμη πέρυσι. Και όμως τη χρειαζόμαστε, γιατί ακούμε για ένα σωρό χημικά δηλητήρια, πραγματικά ενδοκρινικούς διαταράκτες και ένα σωρό άλλες ουσίες, οι οποίες κυκλοφορούν στο περιβάλλον μας και μπαίνουν και στην τροφική αλυσίδα. Αυτή είναι μια τεράστια απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Συμφωνείτε ότι πρόκειται για μια σοβαρή βλάβη στην υγεία μας που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έπειτα η συνεχιζόμενη παρουσία ουσιών σε καθημερινά αντικείμενα που χρησιμοποιούμε και που είναι βλαβερές. Ένα σωρό θέματα, τα ποτήρια, ένα σωρό άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή ε, βάση δεν ε, είναι κάτι σοβαρό και το γεγονός ότι δεν υπάρχει και ισότητα ε, μεταξύ όλων μας, γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν συμμορφωθεί με τις προτάσεις για το REACH, άλλοι όχι και παρόλα αυτά δεν κινδυνεύουν ε, με πρόστιμα. Μια που εσείς είσαστε υπουργό σε μια χώρα που έχετε την υπηρεσία για τα χημικά που φροντίζει για συμμόρφωση, εσείς τι πιστεύετε για όλα αυτά, τα, όλες αυτές τις ουσίες από τις οποίες κινδυνεύει η ανθρώπινη υγεία. Δεν θα έπρεπε η υλοποίηση των μέτρων ε, να επιτευχθεί επιτέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εφαρμογή των μέτρων και συμμόρφωση. Από το, την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία δεν έχω κανέναν. Από το ECR, η Κοψίνσκα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για το πολύ φιλόδοξο αυτό ε, φιλανδικό πρόγραμμα, πρόγραμμα της Φιλανδικής Προεδρίας. Οι προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας ε, μου δημιούργησαν μεγάλο ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, η ισορροπία ε, να υπάρχει. Ε, είναι καλή η προσέγγιση που ακολουθείτε. Τον Ιανουάριο πέρυσι η Κομισιόν μας έκανε μια πρόταση σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των ιατρικών τεχνολογιών με αποτέλεσμα ε, προσδοκόμενο να υπάρχει και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρμόδιων οργανισμών. Τα κράτη-μέλη όμως ανησύχησαν με κάποια από τα στοιχεία αυτής της νομοθεσίας. Παραδείγματο χάρη, κλινικές δοκιμές. Ότι θα πρέπει να δημοσιεύουν τα πορίσματα, να συντάσσονται εκθέσεις. Επίσης, τι γίνεται με την επιστροφή του κόστους θεραπείας. Τα κράτη-μέλη έχουν και άλλους φόβους ε, σε ό,τι αφορά την δυσκολία ε, της εφαρμογής στην πράξη όλων αυτών των διατάξεων. Φέτος το Δεκέμβριο 9 του μήνα θα γίνει μια επόμενη συζήτηση και θα ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή, ε, ε, μάλλον η Προεδρία σας, ώστε να έχουμε μια ικανοποιητική εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα. Ε, e. Ευχαριστούμε. Γκουε, Πάλας. Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ. Ο πόλεμος στα νοικοτικά ήταν αποτυχία. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Έχετε προοδευτική θέση όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Βλέπετε εσείς τους κοινωνικούς κινδύνους όσον αφορά την χρήση τους και θα δουλέψετε για τη διατύπωση μιας νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα νέο πρόγραμμα δράσης, γιατί αυτό που έχουμε, ε, που εκπνέει το 2020, δεν ήταν αρκετά επιτυχές. Έπειτα έχω μια δεύτερη ερώτηση. Απογοητεύτηκα που χτες άκουσα τον Υπουργό για το πώς θα χρησιμοποιείτε το γλυφοσάτ και όχι τόσο για το αν θα εγκριθεί όχι. Όμως το γλυφοσάτ είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να επιτρέπεται κοντά στην διατροφική αλυσίδα. Η ανεξάρτητη επιστήμη έχει δείξει ότι είναι κακό για την υγεία μας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων. Η καλύτερη επιστήμη που μπορεί να αγοράσει η Μονσάντο βέβαια και άλλοι έχουν καταλήξει σε διαφορετικό συμπέρασμα, αλλά εγώ αυτά ε, δεν τα παίρνω της μετρητής. Επίσης κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στο θέμα της ε, ψυχικής υγείας. Και χάρηκα. Εμείς στη χώρα μου στην Ιρλανδία έχουμε πολλά ζητήματα με αυτό το θέμα. Και δυστυχώς η κυβέρνησή μας αλλά και οι προηγούμενες μας έχουν απογοτεύσει πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο έχουν αντιμετωπίσει τα θέματα ψυχικής υγείας και κυρίως τα παιδιά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, δεν θα έπρεπε όλοι μαζί να πιέσετε την Ιρλανδική κυβέρνηση για να κάνει περισσότερο όσον αφορά το θέμα της ψυχικής υγείας. Ευχαριστώ. Πέντε με 7 λεπτά περίπου για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Εξαιρετικές οι ερωτήσεις σας. Πολλές. Θα είμαι σύντομη. Θέλω ξεκινώντας να σας καθησυχάσω, όπως, όπως είπα ήδη. Έχουμε σαφή προσήλωση στη μέγιστη δυνατή πρόοδο και είμαστε διατεθειμένοι να, ε, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ε, των θεμάτων με τρόπο όμως, όπως είπα, ρεαλιστικό και πρακτικό. Ωστόσο, εξαρτόμαστε από τα κράτη-μέλη μπορεί σε σχέση με τις προσδοκίες που έχουμε να αποδειχθούν υπέρογγες οι προσδοκίες. Γι' αυτό λέω ρεαλιστικό και πρακτικό. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε μία διέξοδο για το θέμα των ορμονικών διαταρακτών, χωρίς όμως να μπορώ να υποσχεθώ, όπως πριν κλείσει ο χρόνος θα έχουμε βρει συμβαστική λύση. Η ομάδα μας είναι εξαιρετική. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν για να επιτύχουμε. Μετά είχαμε μια σειρά από Ας ξεκινήσουμε με την αντιβιωτική με την, με την ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά των οργανισμών. Ε, εννοείται ότι ξέρετε πολύ καλά, δεν χρειάζεται εγώ να τονίσω πόσο σημαντικό, σοβαρό θέμα είναι, πόσο μεγάλη απηχή απειλή συνιστά. Και οπωσδήποτε έχει πολύ μεγάλη σημασία η συνεργασία μεταξύ όλων των ε, τομέων για την αντιμετώπιση τη αντιμικροβιακή αντίσταση των οργανισμών. Αλλά αυτό σημαίνει ιδιαίτερω βέβαια και του επαγγελματίε τη υγεία, ε, κτηνιάτρου, ε, παραγωγή, γεωργική και ούτω καθεξής. Πολλά βήματα έχουν υλοποιηθεί. για να ενισχυθεί περισσότερο ο αγώνας αυτός, τον οποίο αποδιόμαστε εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε το πρόγραμμα δράσεως το 2017 το 2018 και επίσης και τελευταία τώρα τον Ιούνιο, 14 Ιούνιου του 2019 με τα συμπερασμάτα του Συμβουλίου για τα προσεχή βήματα ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τις καλύτερες επιδόσεις στην καταπολέμηση της αντιμικροβιακής αντίστασης. Και σε αυτά όλα τα βήματα πιστεύω το Συμβούλιο ε, θέτει το δάκτυλο πάνω στα σωστά ζητήματα πολυτομεακά προγράμματα δράσης, μακροχρόνια, συντονισμό και ε, εποπτεία των μηχανισμών των κρατών μελών και άλλα τέτοια. Επομένως πρέπει να δουλεύουμε εις βάθος, πρέπει να βελτιώσουμε τη διεθνή μας συνεργασία, να εξασφαλίσουμε καλύτερη θέση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη της ε, και κατάσταση αντιμετώπισης της αντιμικροβιακής αντίστασης. Εμβολιασμοί. Πολύ εύστοχα το θέσατε, πιστεύω. Είναι κύριο ζήτημα και στόχος η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Και πολλοί υπουργοί στα κράτη μας ε, αγωνίζονται καθημερινά με στόχο ακριβώς να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνεται με ασφαλή τρόπο εμβολιασμό πάντα, ότι δηλαδή πάντα θα πιστεύει ο πολίτης στον εμβολιασμό. Θα έχει εμπιστοσύνη. Το Δεκέμβριο του 2018 το Συμβούλιο υιοθέτησε σύσταση για το θέμα αυτό που διαπιστώνουμε πως ε, πολλά ακόμα μένουν να γίνουν και κυρίως στην υλοποίηση μετά έχουμε βέβαια την πρόσβαση στα φάρμακα, έχουμε τις ελλείψεις σε εμβόλια που συνιστούν σημαντικές προκλήσεις και μάλιστα σε επίπεδο γενικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο θέμα είναι ότι η αγορά των αντιβιωτικών είναι συγκεντρωμένη, δηλαδή λίγες είναι οι φαρμακευτικές εταιρείε οι οποίες παράγουν το 90% όλων των εμβολίων στον κόσμο. Επομένως έχουμε μεγάλες προκλήσεις, πολλά θέματα, συναφή μεταξύ τους τελικά. Και από αυτά θα εξαρτηθεί και η εμπιστοσύνη του κοινού στα εμβόλια. να δω, το θέμα του καρκίνου. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως ε, συμφωνούν ότι είναι μεγάλη πρόκληση με τη γύρανση του πληθυσμού. Τα ίδια προβλήματα εμφανίζονται όλο και πιο συχνά. Και το θέμα βεβαίως είναι τι μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά, γιατί αυτές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε μεταξύ άλλων. Η κυβέρνηση συνασπισμού στην Φινλανδία έχει μπροστά της μια απέτηση, έχει απέναντι μια απέτηση και να δείξουμε ότι μπορούμε να μεριμνήσουμε, να φροντίσουμε, να προσφέρουμε καλύτερη αγωγή και θεραπεία, αλλά και να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή συνεργασία στο θέμα του καρκίνου. Ψηφιακή υγεία θα είναι το τελευταίο. Το αφήνω για το τέλος. Ξέρετε πως η Φινλανδία επενδύει πολύ στην ψηφιοποίηση έχουμε σημαντική πρόοδο εξασφαλίσει. Πρέπει όμως και να εστιαστούμε στο γεγονός ότι ο πολίτης χρησιμοποιεί υπηρεσίες, τεχνικές συμβούλες που διαρκώς παρακολουθούν την υγεία του. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε περισσότερα ακόμα με τα μοντέλα που έχουμε μέχρι τώρα. Ενώ πρέπει να κάνουμε περισσότερα, χρειάζεται να ανακαλύψουμε νέους τρόπους για το πώς θα το κάνουμε αυτό. Νέους δρόμους με δυναμικό για ε, να καταστεί δυνατή πιο προσωποποιημένη η ιατρική φροντίδα, αλλά και πιο προσιτή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη χρήση των δεδομένων για τη δημόσια υγεία εμείς θεωρούμε στη Φιλανδία ότι μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη νομοθεσία στην ε, δευτεροβάθμια παράγωγη χρήση ε, δεδομένων υγείας ή κοινωνικών δεδομένων που εξασφαλίζουν την καλύτερη χρήση, που θα εξασφαλίσει την καλύτερη χρήση των δεδομένων αυτών για την ε, έρευνα, για την καινοτομία, αλλά και για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνω έκκληση προς εσάς, δεν πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και αυτά είναι μία από τις, μία από τις προκλήσεις στις οποίες θα πιέσουμε για περισσότερη πρόοδο, γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μοιραζόμαστε περισσότερα. Έχουμε καλές πρακτικές στα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να βρούμε και καλύτερα εργαλεία έτσι ώστε και να θεραπεύουμε καλύτερα τους ε, ασθενείς και να ενισχύσουμε το επίπεδα της υγείας και να βοηθήσουμε καλύτερα τον πολίτη στη διαφύλαξη της υγείας του. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σαφή τα μηνύματα. Ξεκάθαρα. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο σε 12 βουλευτές για τον επόμενο γύρο των ερωτήσεων. Εύα Κόπατς, καταρχάς από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω ε, που δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα της δημόσιας υγείας. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Στο πλαίσιο της Φιλανδικής Προεδρίας θα προωθήσετε την αποτελεσματική καταπολέμηση ε, του καρκίνου που είναι ο μεγαλύτερος δολοφόνος του 21ου αιώνα είπατε ε, ότι θα πάρετε βρείτε τις πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό. Θέλουμε να υπάρξει ένα πανευρωπαϊκό αγώνα κατά του καρκίνου και καλό είναι να αξιοποιηθούν σίγουρα οι εμπειρίε όλων των κρατών μέλων. Όλα αυτά όμω απαιτούν χρήματα. Αν θέλουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα μα δώσει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε να λειτουργούν καλύτερα τα εθνικά συστήματα υγεία Και όσο πιο γρήγορα το κάνουμε αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα το καταλάβουν και θα το αντιληφθούν και οι συμπολίτε μας. Ευχαριστώ πολύ. Σάρα Σέρντα από τους ε, Σοσιαλιστέ και Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα. Ακούσαμε που εστιάζει η Φιλανδία σε ό,τι αφορά την υγεία που πρέπει να σωματωθεί σε όλες τις πηγές, διατομεακή προσέγγιση που συστηματικά λαμβάνει υπόψη πώς επηρεάζουν την υγεία οι αποφάσεις ε, και οι δράσεις που λαμβάνονται στο δημόσιο τομέα. Πρόκειται για μια πρόκληση. Και θα το έχει αυτό όπως και το 2006 το επέκεντρο η Φιλανδική Προεδρία. Ελπίζω έτσι να έχουμε καλύτερη υγεία και περισσότερη ευμερία. Ε, πρώτος ε, ε, στις, στους θανάτους είναι οι μεταδοτικές νόσοι. Πάνω από 500.000 πρόοροι θάνατοι. Πρόκειται για 0,8% του ΑΕΠ. Η Προεδρία σας εστιάζει την πρόληψη, την πρωτογενή αυτών των νοσημάτων, ναι ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Βερονίκ ε, Ριγέ Λενουάρ από τη Ρινιού. Κύριε Υπουργέ, ε, θα με συγχωρήσετε που θα επαναλάβω κάτι που υπόθηκε, αλλά είναι μία μείζον πρόκληση. Από καρκίνο πεθαίνουν 1,4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες το χρόνο και 6.000 από αυτούς είναι παιδιά. Έχουμε σίγουρα κάνει πρόοδο με βάση την ανείχνευση, τη διάγνωση και νέα φάρμακα που έχουν ανακαλυφθεί. Αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη σημαντικέ προσπάθειες ε, στον τομέα της πρόληψης της έρευνα, ιδίω ό,τι αφορά την ε, τεχνητή νοημοσύνη, πρόσβαση ε, στην θεραπεία και αντιμετώπιση των προβλημάτων που μένουν μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Ευρωπαϊκό σχέδιο καταπολέμησης ε, του καρκίνου θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ στον αγαπητό πρόεδρο θα πρότεινα μια τροποποίηση του προπολογισμού για να λάβουν υπόψη το ενδεχόμενο ανάγκη χρηματοδότηση. Η Φιλανδική Προεδρία όμω συγκεκριμένα πώ θα υποστηρίξει, ε, πώ θα πλαισιώσει οικονομικά την πρωτοβουλία αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για τους πράσινους ε, η Τίλι Μέτς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας κάνω μια ερώτηση για την ετικετοθεσία σε συσκευασίες τροφίμων. Πολλά έχουν ξεκινήσει να βάζουν κάποιες τέτοιες πληροφορίες διατροφικές εθελοντικά. Και με ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα βλέπουμε ότι αυτό βοηθάει να γίνει σύγκριση της αθρεπτικής αξίας επηρεάζονται επίσης οι επιλογές των καταναλωτών. Πριν από κάποιου μήνε, οι Ευρωπαίοι πολίτε ε, δρομολόγησαν μια πρωτοβουλία, ζητώντας υποχρεωτικά να έχουμε αυτά τα θρεπτικά συστατικά, ε, το θρεπτικό σκορ. Η έκθεση της Κομισιόν ε, θα δημοσιευθεί σύντομα. Πώς θα επιβάλλει τέτοιου είδους συζητήσεις η Φιλανδική Προεδρία, δηλαδή για μια αναρμονισμένη προσέγγιση ώστε να έχουμε απλούστευση της ετικετοθεσίας και των ετροφικών πληροφοριών για να διευκολυνθεί η αγορά και οι καταναλωτές επιλογές τους. Καλή επιτυχία στις επόμενους έξι μήνες. Ωραία. Περνάμε στο ECR για να κονσίσκα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά την ε, αντίσταση στα αντιβιωτικά, που ξέρω ότι ετέθη, αλλά έχω μια πρόσθετη ερώτηση και είναι και σοβαρό το πρόβλημα βέβαια. Ως γιατρός υποστηρίζω κάθε μέτρο πολέμησης της αντίστασης ε, των μικροοργανισμών στα, αντιβιωτικά. Ενώ η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει πως έως το 2050 η μικροοργανισμοί με τη μικροβιακή αντίσταση θα προξενούν τεράστιες ζημιές στη δημόσια υγεία και θα αυξηθούν έως και στα 10 εκατομμύρια το χρόνο ή θάνατοι. Θα ήθελα και μάλιστα εδώ αναφέρομαι στα δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας γιατί ακούσαμε πολλά να λέγονται για ευημερία κοινωνική, οικονομική, εκπαίδευση, όλα αυτά τα βάζετε μέσα. Μια από τις ε, ιδέες λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και καθήκον της, ε, όπως και της Φιλανδικής Προεδρίας, είναι η προαγωγή των μέτρων για τη δημόσια υγεία. Το πρόβλημα των της αντιμικροβιακής αντίστασης δεν είναι ευρωπαϊκό μόνο. Μεταξύ των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν θα έπρεπε να είναι και η κατάρτιση ενός θεματολογίου για τη στενότερη συνεργασία με άλλους οργανισμούς των ανεπτυγμένων κρατών. Πρέπει να αξιοποιήσουμε το υφιστάμενο δυναμικό και γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω τι μέτρα μπορούμε να περιμένουμε από τη Φιλανδική Προεδρία για, τους, ε, για την αντιμικροβιακή αντίσταση. Ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, ένα λεπτό έχετε και επιπλέον μην διαβάζετε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Πρώτον, όσον αφορά την γεωργία. Όσον αφορά τις ενεργές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και που είναι επικίνδυνες και που κυκλοφορούν στην αγορά. Εσείς τι θα κάνετε για να φροντίστε να λυθεί στις χώρες μέλη αυτό το ζήτημα με τις ουσίες αυτές και να είναι πια μια απειλή του παρελθόντος. Δεύτερον, τα υγιεινά τρόφιμα μπορούν να υπάρχουν και μπορούν να αποτελέσουν μια λύση και για την κρίση βιοπικιλότητας και για την προστασία του περιβάλλοντος και μπορούν έτσι να μειωθούν και εκπομπές οξυδίου του άνθρακα. Το κρέας, για παράδειγμα, και η παραγωγή κρέατος είναι υπεύθυνη για περισσότερες εκπομπές οξυδίου του άνθρακα. Εσείς τι θα κάνετε λοιπόν ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια διατροφή πιο υγιεινή όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστούμε. Ελκ Νικολά Εστερλεύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Το θέμα της υγείας των παιδιών μας είναι βασικό. Η υγεία όμως και το μάρκετινγκ που σχετίζονται με τα τρόφιμα δεν βοηθούν. Ρωτώ λοιπόν, σε τι άξονες θα βασιστείτε εσείς για να περιορίσετε τις πρακτικές διαφήμισης που απευθύνονται στα παιδιά με πολύ αλάτι, πολύ ζάχαρη και να καταρρύψετε τους ισχυρισμού ότι κάνουν καλό στην υγεία αυτά τα προϊόντα. Έπειτα, για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλές ε, ουσίες που αποτελούν ε, απειλή για την υγεία μας. Εσείς τι θα κάνετε λοιπόν στην Προεδρία σας, θεσάγετε τα ίδια ε, κριτήρια για τον εντοπισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών όπως κάνετε και για τα λοιπάσματα, για άλλες ουσίες και θα το κάνετε το ίδιο και για τα καλλιτικά και για τα παιχνίδια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σοσιαλιστές. Τίμο Βόλκαν. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα. Η νέα νομοθεσία για τον ιατρικό εξοπλισμό θα ισχύσει από το 2021 χρόνο δηλαδή. Είναι πολύ βασικό να ενισχύσουμε το αριθμιστικό πλαίσιο και να διασφαλίσουμε έτσι την προστασία της υγείας των πολιτών μας, αλλά συγχρόνως να επιτρέψουμε και την πρόσβαση πιο καινοτόμας τεχνολογίας που θα βοηθήσει τις δυνατότητες που έχουμε για την διάγνωση. Το 2019, τον Ιούνιο, η γερμανική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο εξέφρασε ανησυχίες όσον αφορά την βιωσιμότητα και τη δυνατότητα κοινοποίησης ε, νέων ε, ιατρικών εξοπλισμών βάσει του κανονισμού αυτού. Από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν λιγότερα σώματα κοινοποίηση από ό,τι είχαμε κατά το παρελθόν, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολη η κοινοποίηση. Συνεπώ η δικιά σα, η Προεδρία τι θα κάνει για να διασφαλίσει ότι ο κανονισμός για τον ιατρικό εξοπλισμό θα μπορέσει να εφαρμοστεί όπως έχει προβλεφθεί το 2020 και πώς θα φροντίσετε να υπάρχουν αρκετά σώματα κοινοποίηση που να λειτουργούν. Ευχαριστούμε. Ρινιού, παρακαλώ, εσείς πάλι. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Η υγεία των πολιτών σημαίνει καταπολέμηση και των κινδύνων που έχουν να κάνουν με την παρουσία επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον μας και στα προϊόντα που καταναλώνουμε. Εσείς λοιπόν θα πάρετε μέτρα για να διασφαλίσετε την τήρηση του κανονισμού REACH που με τη σειρά του διασφαλίζει την προστασία από επικίνδυνες ουσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τους ενδοκρινικούς διαταράκτες ανά κλάδο. Εσείς θα φροντίσετε η διαδικασία αυτή που έχει καθυστερήσει, δεν θα καθυστερήσει περισσότερο και θα υπάρξει ένα κοινό πλαίσιο για όλους. Έπειτα, κύριε Υπουργέ, μπορείτε να μας πείτε με ποιο τρόπο θα επηρεάσετε τις ευρωπαϊκές πολιτικές στο θέμα του περιβάλλοντος για την προστασία δηλαδή της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών και των παιδιών τους. Ευχαριστώ, Σιντι Φράντσεν, εκ μέρους του ΕΛΚΑ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Υπουργό για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Φιλανδικής Προεδρίας. Καλώς ορίζω την ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται σε μια οικονομία της ευημερία που συνεπάγεται καλή δημοσία υγεία για όλους τους πολίτες. Και αυτό προσφέρει ιδιαίτερη αξία, ιδιαίτερα με την καταπολέμηση, με τον αγώνα για την καταπολέμηση του καρκίνου που γράμισαν και πολλοί συνάδελφοι. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα όμως ότι για να εξασφαλιστεί δημόσια υγεία πρέπει να έχουμε και ένα υγιές περιβάλλον και υπόθηκε και από την κυρία Λάιν ότι θα πρέπει να βρούμε μια στρατηγική η οποία θα προστατεύει τον πολίτη, μια, μια τομεακή, μια ε, οριζόντια στρατηγική η οποία θα προστατεύει τον πολίτη από τη ρήπανση, από τι εκπομπέ, τι βιομηχανικέ από του ενδοκρινικούς διαταράκτε. και επίση έχει καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Συμβούλιο να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα τη δημόσια υγείας, τον περιορισμό των ε, ορμονικών διαταρακτών και να αναλάβει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Ελπίζω λοιπόν η Προεδρία της ε, Φινλανδίας να αναλάβει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή για συνομιλίες μεταξύ Προεδρίας Συμβουλίου, δηλαδή Επιτροπής και Κοινοβουλίου και κυρίως ε, με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσει τον τρόπο ε, προστασίας της υγείας των πολιτών και κυρίως των μικρών παιδιών. Ευχαριστώ. Σχάλτε Μόζαρ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Οι σοσιαλδημοκράτες βλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον ε, και χαρά την μεγάλη προσήλωση που δίνει στα θέματα της δημόσιας υγείας η υπουργό και η Προεδρία. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να αναφερθώ στο θέμα της ε, ατμοσφαιρικής ρήπανσης στην Ευρώπη. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε στα κράτη μας να βελτιωθούν οι τιμές του ατμοσφαιρικού αέρα που αναπνέουμε. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε και κάτι που έθιξαν πολλοί συνάδελφοι οι ε, επικίνδυνες ουσίες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ε, ζωή, ε, ο κάθε πολίτης, πώς μπορούν να απομακρυνθούν από την, τις κοινωνίες μας. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να εμποδιστεί να μπαίνουν στην καθημερινή μας ζωή και γενικότερα το περιβάλλον. Πρέπει να καθαρίσουμε το περιβάλλον από τις ουσίες αυτές. Μια εγγεγραμμένη τώρα. Ο κύριος Κωνσταντίνου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα παρακαλούσα την αξιότιμη κυρία Υπουργό να αναφερθεί κατά τη στη φυλαδική προσέγγιση γύρω από τα ζητήματα της κοινωνικής μέρημνας των προσφύγων και των παρατύπων μεταναστών, ειδικότερα δε γύρω από το ζήτημα της ρεαλιστικής οργάνωσης και λειτουργίας μιας υγειονομική διαδραστικής τους υποστήριξης. Ευχαριστώ. Okay, ε, ευχαριστώ. Ο δεύτερος γύρος λοιπόν ολοκληρώθηκε ως προς τις ερωτήσεις. Πάλι έχουμε κάποια επιπλέον ερωτήματα στην διαδικασία Catch the Eye για την οποία θα δώσω 4 με 5 λεπτά. Δύο συνάδελφοι έχουν στήσει το λόγο από το ΕΛΚΑ. Δύο του ΕΛΚΑ εδώ. Catch the Eye. ECR, πράσινη. Και εσείς ΕΛΚ δεν είσαστε. Όχι, είστε πολύ από το ΕΛΚ. Εκτός και αν ε, δεν ε, προβάλλουν αντιρρήσει οι λοιπέ ομάδες. Ε, θέμα αναλογικότητα όμω Πέτερ, τι. Ας αρχίσουμε λοιπόν αποδεχόμενοι πρώτα δύο αιτήματα από το ΕΛΚΟ. Κύριο Μπουζόη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, εύχομαι πολύ καλή επιτυχία στην Προεδρία σας. Υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με την αντιμικροβιακή αντίσταση, τον καρκίνο. Ε, ήταν πολύ ωραίο το πράγμα που μας δώσατε για τη συνεργασία μεταξύ Φιλανδίας και Εσθονίας, εξαιρετικό. Καλύτερη πρόσβαση στην υγεία λοιπόν, την οποία μάλιστα συστήσαμε και εμείς με τη Ρουμανική Προεδρία και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει περισσότερο στη δική σας Προεδρία. Έχουμε κάποια νομοθετικά θέματα εδώ ανοιχτά. Έχουμε το πρόγραμμα για την υγεία που για πρώτη φορά δεν θα αποκοπεί αλλά θα μπει μέσα σε ένα συνολικό πρόγραμμα. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προτείνει μια μικρή αύξηση στον προπολογισμό που ελπίζουμε ότι θα διατηρηθεί για τις τελικές συζητήσεις. Το HTA, οι ορμονικοί διαταράκτες, ελπίζω, όχι συμφωνώ μάλλον ότι είναι δύσκολο να καταλήξετε συμφωνία, αλλά παρακαλώ βοηθήστε. Είναι εξαιρετική ευκαιρία. Θα ήταν κρίμα για τον Ευρωπαίο ασθενή να μην προχωρήσει το θέμα αυτό. Και επίση πρέπει να γίνει αυτή η αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, δωρεά αίματος ιστών και κυτάρων. Αυτό θα ήθελα να μου πείτε πώς προχωράει σε επίπεδο συμβουλίου. Τι, τι προβλέπετε και κυρία Μονσέρα. Ακούστε. Τρία πράγματα σημαντικά ακούστηκαν. Αντιμετώπιση του προβλήματος του καρκίνου, ψυχική υγεία και αντιμικροβιακή αντοχή. Σίγουρα στα δημόσια συστήματα υγείας υπάρχει πρόοδος, έρευνα, περισσότεροι πόροι και επίσης ε, βοήθεια ε, για τη διάγνωση και τη θεραπεία, ιδίως αυτών των ε, νοσημάτων. Όμως θα πρέπει να εργαστούμε πιο πολύ και να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στην πρόληψη. Πράγματι έχουμε εργαστεί πρόληψη κατά της χρήσης αλκοόλ, ναρκωτικών, διατροφή επίσης. Έχουμε εργαστεί ε, παράδειγμα αρκετά τη καθιστική ζωή, για την εντόπιση παχυσυχή αρκεία κτλ. Όμω, τι κάνουμε σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των συναισθήματων όπω είναι η μοναξιά, το στρε, η κατάθλιψη. Νου υγιή εν τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι, μόν πρόγονοι. Άρα, παρακαλώ, ε, όσο θα έχετε την Προεδρία αυτούς του έξι μήνες, ε, να μας πείτε τι θα κάνετε για να υπάρχει καλύτερη πρόληψη ε, στις, ε, που προανέφερα, αντιμικροβιακή αντοχή, ψυχική υγεία, καρκίνος. Ευχαριστώ πολύ. Χούτα πάλους για τους πράσινους. Σας ευχαριστώ. Μία φιλική επισήμανση. Δεν ξέρω Μήπως δεν το ακούσατε ή δεν το άκουσα εγώ. Αλλά είχα κάνει ερώτημα που δεν μου το απαντήσατε. Και ένα δεύτερο ερώτημα αφορά τις εμπορικές συμφωνίες. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιες φήμες ότι φάρμακα τα οποία έχουν ε, πάρει άδεια ε, στην αμερικανική αγορά μπορούν να έρχονται στην Ευρώπη χωρίς να χρειάζεται να έχουν πάρει προηγουμένως έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Μάλιστα, η Σιάρτα Ιούσκα. Panie Przewodniczący, koleżanki, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις εταιρότητες ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ψυχική υγεία. Είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον το θέμα της εξάρτησης από την ε, κοινωνία της πληροφορίας και το ίντερνετ των νέων μας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Κάνατε λόγο για τους πολέμιους της, ε, ε, των εμβολιασμών. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε νομίζω, από τη βάση, από την αποδοχή και σε αυτό πρέπει να γίνουν και έρευνες για να έχουμε στοιχεία ουσιαστικά και να μπορέσουμε να τα ε, διαδώσουμε. Επιπλέον, πρέπει να καθίσετε σαφές ότι με την αποφυγή των εμβολιασμών υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστούν και να διαχυθούν μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα και κοινωνία ε, μια σειρά από ε, λοιμώξεις. Το άλλο θέμα, το θέμα της δωρεάς αίματος. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και ελπίζω να μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε λοιπόν όλες αυτές τις ερωτήσεις. Έχετε ένα πεντάλεπτο. Άντε, επτάλεπτο για σας. Για τα συμπεράσματα. Ε, αυτό και αν είναι πρόκληση. Να δούμε πώς θα τα καταφέρω να απαντήσω. Ε, χημικές ουσίες στις τροφές. Υπάρχει ένα πληρέστατο πλέγμα νομοθετικό για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν η ΕΦΣΑ, η ΕΚΑ, οι αρμόδιοι δηλαδή αποκεντρωμένοι οργανισμοί που κάνουν εξαιρετική δουλειά στο πεδίο αυτό. Οπωσδήποτε χρειάζεται επιστασία, παρακολούθηση, Έλέγχο της παρουσίας των χημικών, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει η ίδια η αλυσίδα των τροφίμων από το πρώτο βήμα, από την πρωτογενή δηλαδή γεωργική παραγωγή μέχρι την ε, παραγωγή του τελικού προϊόντος να υιοθετήσει ασφαλείς συνθήκες παραγωγής ε, τροφίμων για τους καταναλωτές. Και βεβαίως εμείς, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, όταν έχουμε μπροστά μας τις προκλήσεις είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και σε αυτή να προσαρμοζόμαστε. οι ενδοκρινικοί διαταράκτες. Και είχαμε διάφορες ερωτήσεις πάνω στο θέμα αυτό. Απαντώ λοιπόν ότι η Φιλανδική Προεδρία έχει στόχο να εξασφαλίσει την συμπερίληψη στο πρόγραμμα εργασίας της νέας επιτροπής όλων των μέτρων που θα απαιτηθούν για την αντιμετώπιση των ε, ορμονικών διαταρακτών με σαφή χρονοδιαγράμματα, με φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα. Ο καλύτερος τρόπος είναι να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο για τους... Ε, ε, ο καλύτερο τρόπο για να έχουμε ένα καλύτερο πλαίσιο για τους ορμονικού διαταράκτες είναι να εξασφαλίσουμε ένα στο δυνατόν πιο καθαρό, μη τοξικό περιβάλλον το ταχύτερο δυνατό με βάση βέβαια και το 7ο πρόγραμμα δράσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σήμανση, μάλλον επισήμανση τροφίμων η αναγραφή. Και εδώ είχαμε κάποιες ερωτήσεις, θα πω δύο λόγια. Το Συμβούλιο προσδοκά πως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει την αξιολόγηση των συνεπειών των διαφορετικών ε, νομοθεσιών που έχουν τα κράτη-μέλη ως προς την ε, αναγραφή συστατικών σε τρόφιμα και άρα θα προχωρήσει σε μια ενδεχομένως ε, νέα προσέγγιση, ενδεχομένως για εναρμόνιση ή ένα νέο πλαίσιο νομοθετικό το οποίο εφόσον κατατεθεί θα είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε όσο προλαβαίνουμε. κανονισμός ε, ε, μηχανημάτων ε, και εξοπλισμού ιατρικού. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε στενά. Είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την Επιτροπή, του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου για να βρούμε λύσεις. Και αν καταστεί απαραίτητο, θα δούμε, θα δούμε Πάντως πιστεύω ότι έχουμε πολύ σκληρή δουλειά στο θέμα αυτό μπροστά μας. Ναρκωτικά. Και ζητώ συγγνώμη που δεν το απαντήσα νωρίτερα. Ναι, συμφωνούμε σε μια ολιστική προσέγγιση στο πρόβλημα των ναρκωτικών. Είναι σημαντική Βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη τι συμβαίνει και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να επενδύουμε περισσότερο και στην πρόληψη αλλά και στη σωστή φροντίδα. Τα ναρκωτικά σχετίζονται βέβαια και με τα θέματα της ψυχικής υγείας Και πρέπει να βρούμε κοινού τρόπου συνεργασία στα κράτη-μέλη, μια πολετομιακή δηλαδή προσέγγιση, μια οριζόντια προσέγγιση που χρειάζεται. Για την ψυχική υγεία είχαμε μια ερώτηση. Όπως είπα και νωρίτερα στην ομιλία μου, είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Ευρώπης η ψυχική υγεία, εάν δεν ε, αντιμετωπίσουμε εγκαίρως ε, την πρόκληση αυτή. Θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Έχουμε πολλούς νέους με προβλήματα γιατί δεν έχουν ε, εκπαίδευση, δεν έχουν λάβει εκπαίδευση, δεν έχουν δυνατότητες για απασχόληση. Και εδώ το θέμα δεν είναι η εκπαίδευση, αλλά η ευημερία, γιατί θα μας οδηγήσει σε πολλά άλλα προβλήματα το πρόβλημα αυτό. Οπωσδήποτε λοιπόν θα θεωρήσω ευπρόσδεκτη ή αδίποτε πρωτοβουλία στον τομέα αυτών. το μέλλον ε, της ε, συνεργασίας για την υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν ένα άλλο από τα ερωτήματα. Είναι πολλές προκλήσεις που τις βλέπουμε και οπωσδήποτε πιστεύουμε ότι, ότι η δημόσια υγεία είναι κοινό μέλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού λοιπόν και να το κάνουμε και καλύτερα. Αυτό. Εκεί πρέπει να κοιτάξουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία σε αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω αν λησμόνησα κάτι, εάν σε κάποιον δεν απήντησα. Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν βλέπω να δυσφορεί κανείς. Να, στρατηγική ευημερία της, ε, της Φιλανδικής Προεδρίας. Απαντάτε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, σας καλώ να δουλέψετε και σε σκληρά το δικό σας μετερίζει για να προαγάγετε τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη. Όλοι μας μπορούμε να τα καταφέρουμε μαζί. Έχετε ε, πολλά να προσφέρετε και εσείς. Υποστηρίξτε παρακαλώ το έργο μας. Εμείς υποστηρίζουμε το δικό σας και νομίζω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι να διαπιστώσουμε και τα διακυβεύματα σε περίπτωση που δεν προχωρήσουμε όλοι μαζί. Thank you for... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το συμπέρασμα, αλλά να είσαστε σίγουροι ότι η όρεξη δεν μας λείπει εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε καλά μαζί. Ωραία, θα συνεχίσουμε το, τις εργασίες της Επιτροπής μας σήμερα το απόγευμα στις 5. 5. και θα προεδρεύσω.